Χαίρομαι πάρα πολύ να πω που έφτασε στο τέλος η ακρόαση. Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις ερωτήσεις και για την ευκαιρία που μου δώσατε να εκθέσω τις δικές μου απόψεις. Ίσως ξέρετε πως ε, πυροβατώ, περπατώ πάνω στη φωτιά και υπήρξαν κάποιες φορές που νόμιζα πως θα καώ. Αλλά τελικά νομίζω πως δεν τα κατάφερα. Πως τα, τα κατάφερα. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτά τα πέντε λεπτά για να σας ε, πω ξανά ότι αυτές οι τέσσερις μέρες πραγματικά μου έδωσαν μεγάλη ορμή και με έκαναν να αγαπήσω αυτόν τον τομέα των μεταφορών. Αυτός είναι ένας τομέας ο οποίος επιφέρει ποιότητα ζωή, συνδεσιμότητα και καινοτομία και πιστεύω πως είναι αναγκαία αυτά έτσι ώστε να ευημερούν οι επιχειρήσεις και οι άνθρωποι και η Ευρώπη. Και μπορούμε να πούμε με σιγουριά πως όταν σταματούν οι μεταφορές, σταματούν τα πάντα. Και πραγματικά αυτό δημιουργεί μια τεράστια υποχρέωση, είναι όμως και κάτι συναρπαστικό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τις μεταφορές να έχουν υψηλές επιδόσεις, να είναι σωστά συνδεδεμένες, αξιόπιστες, ασφαλείς και βιώσιμες. Και για να γίνει αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί ο ενιαίος χώρος ευρωπαϊκών μεταφορών. Και μόνο έτσι οι μεταφορές θα συνεισφέρουν στην οικονομική ανάκαψη της Ευρώπης για... και στην ε, ενιαία αγορά. Και πραγματικά αυτός ο στόχος θα είναι η πρώτη μου προτεραιότητα. Όπως ε, άλλωστε αναφέρεται και στις ε, πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου κ. Γιούνκερ. Γνωρίζω τον ζωτικό ρόλο των μεταφορών στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και αναγνωρίζω επίσης πως πρέπει για να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις χρειαζόμαστε ετοιμότητα στις επενδύσεις και στην ε, καινοτομία. Έχω κοινωνικό προσανατολισμό ε, περισσότερο και, γνωρίζω πως ε, χρειάζεται απελευθέρωση έτσι ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα. Ωστόσο πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ό,τι και να κάνουμε ωφελεί τους πολίτες και βελτιώνει τη ζωή μας. Και για μένα αυτό είναι το βασικό. Είμαι λοιπόν δεσμευμένη να παρέχω συγκεκριμένες απαντήσεις στις ε, για υψηλές επιδόσεις στις μεταφορές και ασφάλεια και φιλικότητα προς το περιβάλλον. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής, μπορώ να σας υποσχεθώ ότι όποια πρωτοβουλία και αν αναλάβω θα γίνει με γνώμονα το καλό και το όφελος που θα επιφέρει στην ποιότητα ζωής του Ευρωπαίου πολίτη. Εάν εκλεγώ η επόμενη Επίτροπος Μεταφορών, μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα δώσω στην θέση αυτή καινοτόμο πνεύμα και πάρα πολύ όρεξη και πάθος για δουλειά και για συνεργασία με εσάς, με αυτήν εδώ την Επιτροπή Μεταφορών, διότι πιστεύω ότι όποιο πρόβλημα δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι, εμείς οι ίδιοι μπορούμε και να το λύσουμε. Και αυτό θα γίνει όταν συνεργαστούμε. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε τις ε, μεταφορές να πάρουν πάλι την πρώτη θέση στο πολιτικό θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να κάνουμε τις μεταφορές ραχοκοκαλιά της ε, οικονομίας που χρειάζεται και αξίζει η κοινωνία μας και πως μόνο μαζί μπορούμε να διαμορφώσουμε το μέλλον των ευρωπαϊκών μεταφορών για τα επόμενα πέντε χρόνια. Και σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Also nach Μετά λοιπόν από αυτήν την τελευταία ομιλία της υποψήφιας επιτρόπου φτάνουμε στο τέλος αυτής της ακρόασης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, ευρωβουλευτές, όλα τα μέλη αυτής της Επιτροπής ε, για τις ε, πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις τους και να ευχαριστήσω επίσης και την κυρία Μπούλτς για τις περιστατωμένε απαντήσεις της. Ξέρω πως δεν ήταν εύκολο, πέρασε όμως τώρα. Οι συντονιστές και οι αντιπρόεδροι τώρα θα κληθούν να αξιολογήσουν αύριο το πρωί την ακρόαση της υποψήφιας επιτρόπου στις 8.30 το πρωί στην αίθουσα ΒΙΚ 200 και αυτή η συνεδρίαση θα γίνει και κλεισμένων των θυρών. Και τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς για την δουλειά και την υπομονή τους αυτή την μεγάλη βραδιά. Καταφέραμε μάλιστα να τελειώσουμε και 6 λεπτά πριν και 6 λεπτά νωρίτερα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω και ολοκληρώνεται εδώ η συνεδρίαση.